να τις διαβάσω, μπορείτε να τις εξετάσετε. Μία άλλη πληροφορία. Ε, οι τελικές δικαστικές αρχές ζήτησαν την άρση της ασυλίας του Ευρωβουλευτή Ρομπέρτο Φιόρε, Ιταλού Ευρωβουλευτή, για ένα θέμα που εκκρεμωδικεί στο δικαστήριο της Βιτσέντζας. Με βάση τον κανονισμό, το αίτημα αυτό θα παραπενθεί στη νομική επιτροπή που είναι αρμόδια καθήλια για τα θέματα αυτά. Επίση, η αρμόδια Καθήλια επιτροπή ε, μου έθεσε ένα ερώτημα για ψήφισμα δεύτερης ανάγνωσης που θα συμπεριληφθεί στα πρακτικά της σημερινή συνόδου. Σύμφωνα με το άρθρο 216 του κανονισμού θα θεωρηθούν εγκεκριμένες αυτές οι διατάξεις αν ε, στην ε, γνωστή προθεσμία δεν υποβληθούν προτάσεις ε, για την ε, διεξαγωγή ψηφοφορίας. Αυτές ήταν ε, οι ανακοινώσεις του Προέδρου.